Shall we ε, Να ξεκινήσουμε και αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Είναι το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης για την πρωινή συνεδρίαση. Είναι η παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης για το νέο μέσο γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Είμαι η συγγήτρια της ΛΥΜΠΕ. Αυτή η πρόταση γίνεται στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θέτει τις βασικές προτεραιότητες καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο για την δράση της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και τα προγράμματά της στο εξωτερικό. Ο στόχο είναι να έχουμε ένα μέσο διεθνού συνεργασία, ούτω ώστε να προωθήσουμε τι αξίε τη Ένωση και τα συμφέροντα τη Ένωση σε όλο τον κόσμο. Ούτω ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης με βάση τα όσα πρεσβεύουν οι συνθήκες. Αυτό, είναι που, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ε, Επιτροπή μας είναι το τμήμα της πρότασης καονισμού που μιλάει για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, όπως λέει, στις ανάγκες και στις ευκαιρίες που συνδέονται με τη μετανάστευση λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές τη Ένωση για τη μετανάστευση. Για να συνεισφέρουμε σε αυτό το στόχο, η Κομισιόν προτείνει ότι 10% του ποσού του μέσου να δοθεί για να αντιμετωπίζουμε τις ε, ρίζες της ε, μετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης και της αναγκαστικής ε, μετατόπισης και εκτοπισμού και να διαχειριστούμε και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών, νομίμων μεταναστών, καθώς και προσφύγων στα πλαίσια του κανονισμού. Και τώρα θα πάρω το λόγο και συνεχεία θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Δεν βλέπω κανέναν. Κρίμα είναι. Α, έχει έναν. Τέλεια, ευτυχώς. Έχει ένα σκιώδη εισηγητή. Θα μιλήσω Ιταλικά, γιατί προετοίμασα την παρέμβασή μου στη μητρική μου γλώσσα. Το καθήκον μας είναι να τροποποιήσουμε την πρόταση από τη σκοπιά της ΛΥΜΠΕ. Αυτό προσπάθησα να κάνω, παρότι είναι δύσκολη η προσπάθεια αυτή, γιατί πολλά ε, θέματα ε, έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη ΛΥΜΠΕ, αλλά χωρίς να είναι η ΛΥΜΠΕ καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Θα εστιάσω σε τρεις τομείς που είναι βασικοί για μας και υπάρχουν στην γνωμοδότησή μας. Θέλω να εκφράσω εγνωμοσύνη καταρχά στου κοιόδη ηγητέ, παρότι δεν υπάρχουν, δεν είναι εδώ μέσα, για τη συνεισφορά και την συνεργασία του. Πολύ σύντομα, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα τρία σημεία. Ο πρώτο τομέα είναι ο τομέα τη μετανάστευση. Οι τροπολογίε που προτείνω γι' αυτό έχουν σαν σκοπό να μην αφαιρέσουμε ποσά από το βασικό πεδίο εφαρμογή τη πρόταση, δηλαδή από του στόχου που απαριθμεί το άρθρο 3 Κατά την άποψή μου, λείπει στον κατάλογο των στόχων μία σαφής αναφορά στην, ε, στο θεματολόγιο 2030, στην καταπολέμηση της στόχιας, της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της ανισότητας. Αλλά βεβαίως αυτό δεν είναι θέμα δικής μας αρμοδιότητας. Ο κανονισμός σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που συνδέονται με την ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν θα έπρεπε με άλλα λόγια να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για στόχους βραχυπρόθεσμους της ε, εξωτερικής πολιτικής ή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος τομέας αφορά το νομικό πλαίσιο. Η πρόταση παρουσιάζεται λίγο ελλειπτική, έχει κάποια κενά από αυτή την άποψη. Πιστεύω θα ήταν κρίσιμο και σκόπιμο να αναφέρουμε πολύ ρητά, πολύ συγκεκριμένα τους ευρωπαϊκούς ε, κανόνες και διεθνεί κανόνες ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ε, που αφορούν τη διατήρηση της γης. Όπως τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, τη Δήλωση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Τρίτον, και τελευταίο στοιχείο, τελευταίο τομέα, η governance, η διαχείριση δηλαδή του μέσου αυτού. Κάποιες τροπολογίες που σας προτείνω δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ρόλο θεματοφύλακα. Η Κομισιόν θα έπρεπε να κληθεί να υποβάλει στους Ευρωβουλευτές μια ετήσια έκθεση για τα ποσά που χορηγούνται. Επίσης, πάντα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αποκατασταθεί ο μηχανισμός ε, που λέγεται Grievances Mechanism, ε, μηχανισμός δηλαδή παραπώνων, που, που προβλέπεται από το Μηχανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά δεν προτείνεται στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus, συν. Όλοι που ενδιαφέρονται για τα project που χρηματοδοτεί το νέο μέσο, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν παράπονα και αμφισβητήσει στην Κομισιόν. Επίση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν συχνά επί τόπου. Να τον αναγνωρίσουμε όταν προωθούν την ε, κοινωνική ανάπτυξη και την καταπολέμηση τη φτώχεια. Η πρόταση τροπολογία είναι αυτέ οι οργανώσει να δίνουν τη γνώμη του συστηματικά, να τι διαβουλευόμαστε ε, συστηματικά, ούτω ώστε να παίρνουμε αποφάσεις πιο κοντά στις ανάγκες τους στις ανάγκες για ενίσχυση των πιο αδύναμων, με μια ειδική έμφαση στις γυναίκες, στα παιδιά και στους ανηλίκους εν γέννη. Σας ευχαριστώ και σας ρωτώ αν έχετε ερωτήσεις ε, ή αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά. Um, Ευχαριστώ. Ω κοιόδης συζητητής ε, της ομάδας CCR, καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν, δήμα προς την κατεύθυνση, είναι λίγο ο κ. Βίστησεν, για να εφαρμοστεί αυτό το μέσο διεθνούς συνεργασίας, γειτονίας και ανάπτυξης. Ε, οι περισσότερες πρωτοβουλίες της Κομισιόν είναι προς κατεύθυνση. Θα θέλατε ίσως να είναι πιο φιλόδοξη η πρόταση της Κομισιόν, αλλά αυτό θα εξασφαλιστεί χάρη στις τροπολογίες που θα περάσουμε για αυτή την γνωμοδότηση. Επίσης, ε, διέτρεξα το σχέδιο γνωμοδότησης της ηγητρίας. Η άποψή μας είναι ότι έχουμε αρκετές διαφορές απόψεων. Γι' αυτό λοιπόν θα υποβάλουμε τη δική μας γνωμοδότηση και θα δούμε που θα πάει το πράγμα. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, γνωμοδότησή σας που θεωρώ ότι κινείται προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο θέλω να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με την ε, γνωμοδότησή σας. Διαπιστώνουμε ότι το NDSCI ε, εντάσσεται στο, στο πλαίσιο των ε, στόχων για το 2030, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ίσως αυτό δεν αναδεικνύεται επαρκώς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει η διαδικασία αυτή να ε, υπαχθεί στη συνολική διαδικασία της ε, ατζέντα για το 2030. Η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους ε, υπάρχει, πρέπει να, να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπατε, το μέσο αυτό έχει ως στόχο την εξάλληψη των ε, ριζικών αιτίων της ε, μετανάστευσης και σε αυτό το, σε αυτό το τομέα περιλαμβάνονται δράσεις όπως είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων που υποστηρίζονται βεβαίως από την Κομισιόν όμως είναι σημαντικό να συγχωνεύσουμε, να συνδυάσουμε την αναπτυξιακή με την μεταναστευτική πολιτική. Επίσης, χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας και την ε, παραπομπή σας στις ε, διεθνείς ε, δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαρά μας να εντάξουμε αυτές τις αναφορές και στο κείμενο, αν και εμείς θεωρούσαμε ότι έτσι κι αλλιώς εξυπακούεται, αλλά καθόλου βεβαίως δεν θα έβλαπτε, όπως προτείνετε εσείς, να υπάρχει και ρητή αναφορά. Για την έκθεση FSD, να σας πω ότι αυτό που προτείνεται περιλαμβάνεται ήδη στον δημοσιονομικό κανονισμό. Η διαφορά ανάμεσα στο παλιό EFSD και το νέο προτινόμενο EFSD η διαφορά μεταξύ των δύο κανονισμών οφείλεται ακριβώς σε αυτόν τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ και πολλές από τις υποχρεώσεις υπό το EFSD ε, καλύπτονται πλέον από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Γι' αυτό και θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκτελούνται οι ίδιες διαδικασίες δύο φορές. Χαιρετίζουμε και την προσήλωσή σας ε, στην ε, εμπλοκή της ε, κοινωνίας των πολιτών. Συμφωνούμε και εμείς ότι κατά τη χάραξη, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και στο NDACI θεωρούμε ότι και αυτή η διάσταση έχει ενισχυθεί. Υπάρχει διαβούλευση με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις φάσεις, σε όλα τα στάδια και θεωρούμε ότι ε, το NDSDI θα συμβάλλει ακριβώς στην εξάλληψη, στην άρση μάλλον του κατακαιρματισμού των διαφόρων μέσων που υπάρχουν σήμερα μέσω της ε, θέσπισης ενός σαφούς και ενιαίου συνόλου κανόνων. Ευχαριστώ. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε κύριε Σαντεμετέριο για τις εξηγήσει και τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Ελπίζω ότι θα έχουμε και στο μέλλον τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Λοιπόν, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η 6η Νοεμβρίου 5 απογευματινή. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Κλείνω τη συνεδρίαση. Σωστά.